στο Νεπάλ ο αριθμός των θυμάτων έχει πλησιάσει τις 4.000 αυτή τη στιγμή. Πάνω από 6.500 άτομα είναι τραυματισμένα. Έχετε δει όλες τις εικόνες της καταστροφής του Ολέθρου στο Νεπάλ. Βλέπετε τα κτίρια τα οποία έχουν καταστραφεί, έχουν καταρρεύσει, τους δρόμους οι οποίοι είναι πλέον αδιάβατοι ιστορικά μνημεία τα οποία έχουν καταστραφεί, νοσοκομεία τα οποία είναι υπερφορτωμένα, δεν υπάρχει ρεύμα και υπάρχει έλλειψη πόσιμου ύδατος και τροφίμων. Και είναι και ο χειρότερος σεισμός στα Ιμαλάια εδώ και 100 χρόνια. 100.000 παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν, βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση και χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει τα άμεσα ε, μέτρα τα οποία ελήφθησαν για ανακούφιση των θυμάτων από κράτη-μέλη και επίση κάνει μια έκκληση και στου διεθνεί οργανισμού στο ταχύτερο δυνατό να έρθει η βοήθεια στα άτομα τα οποία χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Οι σκέψει μα είναι με τα θύματα του σεισμού και θέλουμε να εκφράσουμε την ε, αλληλεγγύη μα με το λαό του Νεπάλ που επλήγει από αυτόν τον τρομερό σεισμό. Επίση, κυρίε και κύριοι, πριν από μία εβδομάδα εκτελήχθηκε πάλι μια τρομερή καταστροφή στη Μεσόγειο. Μεταξύ 800 και 1000 ατόμων έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη θαλάσσια καταστροφή. Ήταν να διασχίσουν τη Μεσόγειο καταδιωκόμενοι από τον πόλεμο, από την καταδίωξη, από την πείνα, την ένδια για να βρούνε λύσεις στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε πια να κάνουμε κάθε φορά ενό λεπτού σιγή σε κάθε συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπουμε και νιώθουμε ότι κάθε φορά που θυμόμαστε τα θύματα αυτά, τίποτα δεν αλλάζει στην πραγματικότητα. Τίποτα δεν αλλάζει από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να αποτραπούν αυτές οι ανθρώπινες καταστροφές. Και στην τελευταία ολιομέλεια το είχα τονίσει αυτό, και θα έχουμε και σε αυτή τη Σύνοδο μια πλήρη συζήτηση για το θέμα αυτό, τόνισα πόσο μας έχει συγκλονίσει αυτό το οποίο έχει λάβει χώρα. Είχα πει στην προηγούμενη Ολομέλεια ότι ήμουν συγκλονισμένο από το δράμα των 350 θυμάτων, αλλά είχα πει ότι δεν ήλπιζα στην επόμενη Ολομέλεια να μην χρειαστεί να το επαναλάβω αυτό. Την, ε, το λεπτό συγγύηση ή την υπενθύμηση των θυμάτων στην Μεσόγειο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα όλα αυτά. Λόγω της δραματικής λοιπόν αυτής κατάστασης θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι είναι ένα πράγματι θλιβερό γεγονός, ένα γεγονός που μας εξοργίζει από την έλλειψη μέρημνας για τα άτομα που χάνουν τη ζωή της. Και πάλι λοιπόν για τα θύματα του Νεπάλ και για αυτούς που έχασαν της, ε, της ζωής της Μεσογείου. Σας ζητώ να κρατήσετε λεπτό λεπτού Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σταθώ και σε ένα σημείο σχετικά με το οποίο έχουν ε, αναφερθεί πολλοί